Good morning, colleagues. Καλημέρα συνάδελφοι. Αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του φετινού έτους. Σας εύχομαι καλή χρονιά για το 2020 με χαρές και επιτυχίες. Γεμάτη προκλήσεις ήταν αυτή η χρονιά, πολλή δουλειά για την Επιτροπή μας. Ελπίζω να είμαστε επιτυχείς στις προσπάθειές μας. Ως συνήθως ε, έχουμε web streaming, έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 4ης Δεκεμβρίου έχουν σταλεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε με email στις 14 ε, Ιανουαρίου του 2020. Θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης 4 και 5 Δεκεμβρίου του 2019, αν όλοι συμφωνούν. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στην ψηφοφορία. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για την, ε, τον, κανονισμό, τον εκλεκτικό κανονισμό της Κομισιόν που τροποποιεί τον κανονισμό 347 του 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον κατάλογο της Ένωσης για έργα κοινού συμφέροντος ή ενδιαφέροντος καλύτερα. Έχουμε μία αντίρρηση. Όχι... Έχουμε λοιπόν πρόταση ψηφίσματος που φέρνει αντίρρηση ε, σε κατεξιδότηση πράξη σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 111. Ε, το αίτημα Τη Ήτρε για να υποψηφίσουμε για την απόρριψη ε, της πράξη πράξης έχει, που θεσπίζει τον τέταρτο κατάλογο μάλλον, έχει υποσταλεί πάνω από 8 βουλευτές, από δύο τουλάχιστον πολιτικές ομάδες. Να σας ψηφίσω. Εάν ψηφίσετε ναι, ψηφίστε ναι για το, την πρόταση ψηφίσματος που απορρίπτει τον κατάλογο, όχι για, την, για τον κατάλογο. Αν υποστηρίζετε λοιπόν τον κατάλογο, θα πρέπει να απορρίψετε την πρόταση ψηφίσματος. Είναι ακριβώς το ανάποδο, έτσι. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε να γίνει στον κατάλογο. Ας κάνουμε μια δοκιμή ψηφοφορίας. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πρώτη φορά εγώ οργανώνω ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Είναι η πρώτη μου, η παρθενική. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία όλα. Αν είσαστε έτοιμοι, σας καλώ να ψηφίσετε υπέρ κατά του ψηφίσματος που φέρνει αντίρρηση στην κατεξιδότηση πράξη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πολύ ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Να δείξουμε το αποτέλεσμα στην οθόνη. 73 ψήφισαν, 17 υπέρ, 54 κατά, 2 αποχές. Η πρόταση ψηφίσματος ε, για την αντίρρηση δεν περνάει, άρα ο κατάλληλος θα εξακολουθήσει να ισχύει. Πάμε στην πρώτη συζήτηση. Τώρα, οι συνάδελφοι που ήρθαν ειδικά για να ψηφίσουν μόνο, έχουν δύο λεπτά για να αποχωρήσουν. Να πάνε σε άλλες ε, επιτροπές ή σε άλλες συνεδριάσεις. Δύο λεπτά ξαναρχίζουμε τη δική μας συνεδρίαση. Okay, colleagues, uh, let's... Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο σημαντικές συζητήσεις πριν το μεσημερινό διάλειμμα. Το επόμενο σημείο, το 6, είναι μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς έγγραφο για την πλήρη ευρωπαϊκή και συνολική ευρωπαϊκή προσοχή προσέγγιση στην ε, αποθήκευση ενέργειας, αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με τίτλο «Μια σφαιρική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενεργειακή αποθήκευση». Είναι σημαντική η αποθήκευση αυτή για, ένα, για μια ε, καλή ενεργειακή μετάβαση. Η συμμετοχή και η ένταξη των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια απαιτεί ε, λύσει για αποθήκευση ενέργεια. Ο εισηγητής θα παρουσιάσει, ή η εισηγήτρια θα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη για το σχέδιο έκθεση και θα γίνει μια ανταλλαγή απόψε με του και εισηγητές και του υπόλοιπου ευρωβουλευτέ. Έχουμε 55 λεφτά. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κλάουδια Γκαμών. Ζητάω από όλους τους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα να σοπάσουν και να είναι προσεκτικοί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ για να δουλέψουμε πάνω σε ένα κοινό ε, στόχο που είναι να έχουμε μια ε, ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς, προς το διοξείδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, η ζήτηση θα διπλασιαστεί και θα πρέπει να καλύπτεται και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε λοιπόν όμως μια κακή ε, επιρροή ότι θα πρέπει ένα κακό, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, επειδή υπάρχει αστάθεια λόγω των ανανεώσιμων, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό και να εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια του ανεφοδιασμού σε ενέργεια. Και περνάω στο σημαντικό σημερινό θέμα για να έχουμε ουδε κλιματική ουδετερότητα, ε, μετάβαση προς τις ανανεώσιμες και ενεργειακή ασφάλεια. Για να τα κάνουμε αυτά και τα τρία, θέλουμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια. Ε, πρέπει να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι τόσο σημαντικό όσο η παραγωγή ενέργειας και τόσο σημαντικό όσο το έξυπνο δίκτυο. Όταν συγκρίνουμε το δυναμικό των διαφορών τεχνολογικών που έχουμε για την αποθήκευση, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και το αποτύπωμα του άνθρακα. Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική ανάλυση και μια ουδέτερη προσέγγιση απέναντι στις τεχνολογίες. Είμαι πεπισμένη, λοιπόν, ότι πρέπει να κοιτάξουμε κάθε τεχνολογία και να δούμε το ρόλο που μπορούν να παίξουν στο μέλλον. Και η ιδέα τη έκθεση είναι να κοιτάξουμε τι διάφορε διαθέσιμε τεχνολογίε ε, που έχουμε φτάσει, τι χρειάζεται ε, για να τι εκμεταλλευτούμε πλήρω. Και μια και είμαι Αυστριακή θα, ζητήσω, θα ξεκινήσω με την αποθήκευση με αντλίε. Έχουμε ευελιξία και μεγάλο δυναμικό για το δίκτυο. Ε, καλύπτει το 97% της σημερινής δυνατότητας αποθήκευσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία για το πόσο μεγάλο είναι το υπολείπον δυναμικό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το δυναμικό που υπάρχει όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσουμε τις ε, προτεραιότητες. Φερρυπίν, μπορείτε να σκεφτείτε πώς ε, τα έργα αποθήκευσης ε, μπορούν να αναγνωριστούν για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον για να βρούμε την ισορροπία, για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας. Κάποιοι ερευνητέ λένε ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αναβάθμιση των ε, σημερινών εγκαταστάσεων ε, με, νέα φράγματα κτλ. Ε, και αναβάθμιση των παλιών ε, φραγμάτων. Επίσης, ε, δεύτερη τεχνολογία, έχουμε εποχιακή αποθήκευση, δεν χάνουμε την ε, ενέργεια με τη μεταφορά, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή αναρμόνιση για τα ελάχιστα ε, πρότυπα, καθώς και ανάμειξη πηγών. Επίσης, ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, γιατί δεν είναι αποτελεσματική 100% αυτή η τεχνολογία. θα πρέπει να δούμε και τη σταθερότητα των δικτύων. Ε, επίσης, οι τιμές ε, για την παραγωγή εξαρτάται από το εξωτερικό, εξαρ... ανάλογα με το τι είδους ε, ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται και μερικές φορές μπορεί να είναι μεγάλο το αποτύπωμα του, άνθρα, του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την εξάρτηση από εισαγωγές πρώτων υλών, παραδείγματο χάρη να έχουμε μια, ένα κυκλικό σχεδιασμό. Θα πρέπει ε, να γίνεται η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να δούμε τι θα κάνουμε τις μπαταρίες. Ε, γι' αυτό χρειάζεται συνεχής δράση για τις μπαταρίες. Ε, επίσης, ε, υπάρχει ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία με νομοθεσία της Κομισιόν για τις μπαταρίες. Ε, ανάλυση του κύκλου ζωής ε, για το αποτύπωμά του διοξιδίου του άνθρακα και θα πρέπει να δούμε και το δυναμικό που έχουν οι μπαταρίε ε, στα νοικοκυριά με έξυπνη φόρτωση και να χρησιμοποιούμε όλε τι μπαταρίε για να αποθηκεύουμε την ενέργεια. Το φωτοβολταϊκό τόξο. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε τι κάνουμε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ε, ε, ε, θερμοαποθήκευση, ε, αντλίες θέρμανσης. Ε, ε, υπάρχουν ε, επίσης ενδιαφέροντα προγράμματα που χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια και την αξιοποιούν. Θα πρέπει να δούμε το ρόλο που έχουν οι καταναλωτές ευελιξία ε, σε αποθήκευση σε νοικοκυριά με ηλεκτρονικά οχήματα, μπαταρίες. Ε, υπάρχουν ε, ήδη στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια κάποια προγράμματα και πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα. Ε, τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι κάποιοι κανονιστικοί φραγμοί που υπάρχουν ακόμα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη διπλή χρέωση και τη διπλή φορολογία σε ορισμένες χώρες για την ε, λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, κατανάλωση, αλλά και, παραγωγή, το θέμα της παραγωγής. Α, αναθεώρηση του κανονισμού 10E, διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ε, κλιματικοί στόχοι βιωσιμότητας που δεν υπάρχουν ακόμα, ε, δεν έχουν συσσωματωθεί στα project και θα πρέπει να συσσωματωθούν. Ε, επίσης, ε, η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων κοινού συμφέροντος θα πρέπει να εξεταστεί. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υπήρχε ανάπτυξη, έλλειψη μάλλον στα προγραμμάτων ενέργειας στον ορίζοντα 2020 γιατί ε, εστιάζει κυρίως σε δραστηριότητες που είναι πολύ κοντά στην αγορά. Αυτές είναι οι σκέψεις μου για το θέμα αυτό, που θα βρείτε τελικά και στην έκθεση. Θέλω να ακούσω τώρα τις ε, ιδέες σας, γιατί θέλω να τις λάβω υπόψη μου όταν ε, γράψω το κείμενο. Είναι ενδιαφέρον το θέμα, θα είναι η συζήτηση και χαίρομαι που νωρίς νωρίς ασχολείται με το θέμα αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάμον για την παρουσίασή σας και για την έκθεση. Καλή τύχη λοιπόν. Όπως είπατε είναι πολύ σημαντικά τα επιχειρήματα αυτά. Θα περάσω τώρα στους κοιόδες εισηγητές από την κάθε πολιτική ομάδα και θα σας παρακαλέσω να μείνετε στα δύο λεπτά ομιλίας. Η κυρία Σπυράκη έχει το λόγο εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ε, ασαφή φράση, το πεδίο εφαρμογή δηλαδή τη έκθεση. Ε, πολύ φοβάμαι πω η συγκήτρια δεν μα έστειλε αρκετέ πληροφορίε, διότι το θέμα είναι αρκετά ευρύ και θα έπρεπε να καθορίσουμε τις, ε, τους στόχους μας, να δούμε τι θέλουμε από αυτή την έκθεση. Και θεωρώ πως θα πρέπει να εστιάσουμε στις ρυθμιστικές και νομικές προκλήσεις, καθώς και την ορατότητα όλων των project. η τεχνολογία αυτή αναμένεται να διευρυνθεί και θα πρέπει να φροντίσουμε να ενσωματωθεί στο ε, δίκτυο ενέργειας καθώς και να προβλεφθούν δυνατότητες αποθήκευσης. Είναι πολύ βασική για να παρέχει ε, ισορροπία στο σύστημα και ε, να βοηθήσει στην αποκέντρωση του συστήματος ηλεκτροδότησης και στην ενεργειακή ασφάλεια θα δώσει ευελιξία στις επόμενες γενιές και θα συνεισφέρει στη μελλοντική ανάπτυξη. Η αποθήκευση ενέργειας θα βοηθήσει επίσης την αποδέσμευση από άνθρακα των άλλων τομέων και θα βοηθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση τους ε, στην ηλεκτροδότηση κτηρίων, για παράδειγμα. Ε, οι μπαταρίες δεν είναι ικανές να αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα το υδρογόνο μπορεί να ε, μπορεί να αποθηκευτεί σε μεγάλες ποσότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, το υδρογόνο, όταν παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών. Η αποθήκευση ενέργειας δεν, δεν μπορεί να ε, αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τομέα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές πηγές ενέργειας και να σας υπενθυμίσω ότι οι τρεις πυλώνες είναι, είναι πολύ σημαντικοί. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην αγορά να ε, διαχειριστεί την ε, ζήτηση και την προσφορά, να ε, διαχειριστεί την αποθήκευση και να δώσει έμφαση στις ανανεώσιμες. Η οδηγία επίσης προβλέπει δυνατότητες αποθήκευσης μέσω διαφορών διατάξεων. Ωστόσο, χρειάζεται να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ του υδρογόνου αερίου και, της, ε, και του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Κομισιό να παρουσιάσει μία πρόταση στην Ένωση των Διαφορών Τομέων στο πλαίσιο του κανονισμού του κανονισμού και να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΕΝ δεν είναι επιλέξιμη αποθήκευση ενέργειας για χρηματοδότηση παρά μόνο για επιχορηγήσεις. Επίσης πρέπει να αυξηθεί η ορατότητα των ε, project αυτών γι' αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να βοηθήσει μέσω κανόνων την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών και ε, να προτείνει ένα δεσμευτικό όριο για την, τον ε, τομέα. Αυτά καταλαβαίνω από την πρώτη ανάγνωση της ε, εκθέσης της εισηγήτριας και να ξαναπώ ότι δεν λάβαμε ούτε ένα email από εκείνη έτσι ώστε να ξεκινήσουμε δουλειά σε αυτό το project. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σπυράκη. Ο Νίλς Φούγκλισάνγκ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια εξαιρετική ανάπτυξη ε, και εξέλιξη σε ό,τι αφορά τι ε, τιμέ ε, των ανάσχομων πηγών ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά και οι αναμογεννήτριε έχουν πέσει πολύ από πλευρά κόστου, το οποίο είναι θετικό αν θέλουμε να προωθήσουμε τον τομέα των ΑΠΕ για να προωθήσουμε και το στόχο τη καταπολέμησης τη κλιματική αλλαγή. Η μεγάλη πρόκληση όμω είναι ακριβώ το θέμα αυτή τη έκθεση η αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν γίνεται να έχουμε χαμηλή ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, όταν έχουμε απώλεια ε, θερμότητας από τα πορτοπαράθυρα ε, και ούτω καθεξής. Πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λοιπόν αυτό, πώς θα αποθηκεύουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέσσερις ε, τρόπους έχω βρει εγώ τουλάχιστον ε, για την αποθήκευση. Πρώτον, συσσωρευτές έχουμε, βρει, έχουμε δει τρομερή ε, ανάπτυξη της ε, ζήτησης τα τελευταία χρόνια και μπορούμε να δούμε πώς θα την αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη ζήτηση. Δεύτερον, έχουμε ηλεκτροχημική, ηλεκτροχημική ε, αποθήκευση, power to X, όταν χρησιμοποιούμε την ενέργεια για την αποθήκευση του υδρογόνου. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διερευνήσουμε περισσότερο. Θερμική αποθήκευση που ανέφερε η συγκήτρια όταν θερμαίνεται ένα υλικό, για παράδειγμα, το νερό. Και τέταρτον, μηχανική αποθήκευση, όταν ε, ε, ένα αντικείμενο ε, τίθεται σε κίνηση. Ένας τροχός, για παράδειγμα. Όλες αυτές τις άγουσες πρέπει να διαρευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να καταρτήσουμε μια στρατηγική για το πώς θα διοχετεύσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ανέφερε και η συγκήτρια, μίλησε για τον κανονισμό ε, TEN-E, διευρωπαϊκών δικτύων και, τον, ε, και το πρόγραμμα Horizon. Αυτές οι τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας. Πρέπει να κατευθύνουμε λοιπόν κονδύλια του ορίζοντα προς τα εκεί. Προσβλέπω ε, σε αγαστή συνεργασία με την εισηγήτρια για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νενίστο από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την πολύ καλή παρουσίαση του θέματος. Το θέμα της αποθήκευσης θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο της, ε, του γενικότερου συστήματός μας ε, με το πλαίσιο της απομάκρυνσης από τον άνθρακα και να δούμε πώς μπορεί να μας διευκολύνει αυτή η αποθήκευση στην ε, ενεργειακή μας μετάβαση. Θέλουμε ένα σφαιρικό, μια σφαιρική προσέγγιση εφιούς συστήματος και όχι να επικεντρωνόμαστε μόνο στα επιμέρους ε, στοιχεία του, θέλω να το βλέπουμε σφαιρικά για να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και η ενεργειακή αποθήκευση εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Καθώ θα πηγαίνουμε προ ένα σύστημα με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, να δούμε πώ από κλιματική άποψη θα είμαστε φιλόδοξοι ε, και αποτελεσματικοί. Θα ήθελα να θίξω πιο συγκεκριμένα την αποθήκευση τη ε, ψήξη και θέρμανση πάντα με γνώμονα της ΑΠΕ. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει εδώ απομάκρυνση από τον άνθρακα στο Ελσίνκι. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν ε, υπόγειες υποδομές ε, αποθήκευσης και με διάφορες λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θέρμανση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην αποθήκευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαρευνήσουμε. για την θέρμανση των ε, περιοχών. Μετά, ε, να δούμε την ε, ευελιξία των ανεμογεννητριών. Είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει στην Σουηδία και στη Δανία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κάτι άλλο πρέπει να δούμε είναι η αρχή της αποτελεσματικότητας πάνω απ' όλα. Κάποιες τεχνολογίες έχουν σημαντικές απώλειες. 30-40% ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, ε, στις ε, αντιλίες λέμε ότι τα πάνε καλύτερα από τους ερευτές. Αυτό πρέπει να το δούμε. Κάθε φορά πρέπει να εξετάζουμε ποια λύση είναι πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική. Είναι σημαντικός ο φάκελος και θέλουμε να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σίλβια Λιμάρα από την ομάδα ID. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μείνω στα δύο λεπτά. Επί της αρχής θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καλωσορίζω και όλα στο γεγονό ότι γίνεται συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας. Είναι νομίζω θεμελιώδες ε, και πολύ βασικό θέμα. Έχουμε προσπαθήσει λοιπόν ε, να κάνουμε αυτή την έκθεση και ε, ακούω την εισηγήτρια να λέει ότι η αποθήκευση ενέργειας έχει να κάνει με την ευελιξία. Το θεωρώ λάθος αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω πως δεν υπάρχει καμία ευελιξία στην αποθήκευση ενέργειας. Ε, το έχουμε δώσει άλλο όνομα και αυτό λέγεται ενεργειακή ασφάλεια. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι άκουσα από πολλούς πως η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες μορφές ενέργειας, αλλά νομίζω πως έτσι θα χάσουμε χρόνο. Θεωρώ πως ε, οι πολιτικοί θα έπρεπε να αναγνωρίσουν ε, την ε, πρόοδο της τεχνολογίας. Νομίζω όμως πως αν η τεχνολογία ήταν όντως τόσο πρωτοποριακή θα το είχαμε δει να εφαρμόζεται στην πράξη θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλες ε, μορφές ε, παροχής ενέργειας. Η τηλεθέρμανση είναι ε, μια μορφή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στη Φιλανδία, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε μέρους που μπορεί να μην επιτρέπουν την χρήση του, της ίδιας μορφής θέρμανσης. Θέλουμε να είναι κλιματικά ουδέτερη η ε, ενέργεια. Όμως θα πρέπει πρώτα να λύσουμε το θέμα της αποθήκευσης και θεωρώ ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο είναι να βάλει το πίσω πόδι ε, πιο μπροστά, να κάνει παραπάνω βήματα από αυτά που ε, αντέχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Από το ECR ο κύριος Κρασνοντεύσκη, αντιπρόεδρος μας και συντονιστής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια. Πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση της πρωτοβουλία. Ε, γνωρίζουμε όλοι ότι ε, προκειμένου να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στην ενεργειακή αποθήκευση. Και προς αυτό τον στόχο θα πρέπει να έχουμε και ένα κατάλληλο έγγραφο. όπου θα συγκεντρώνονται τα βασικά ζητήματα. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το θέμα των συσσωρευτών και των υπολείπων ε, τεχνολογιών. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπει στην αγορά παραγωγής συσσωρευτών ε, στη δεύτερη γραμμή, αν θέλετε. Ε, λίθιου, μπαταρίες λιθίου και λιθίου. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε το κόστος ε, παραγωγής ε, για τις πρώτες ύλε. Ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό από την Ασία. Να δούμε λοιπόν νέες τεχνολογίες που αναμένεται να υπάρξει πολύ σημαντική εξέλιξη στο μέλλον για το υδρογόνο, ε, παράγωγα χημικά και το καθεξής, προκειμένου και η Ευρώπη στο τέλος να έχει ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Μετά, οι φραγμοί που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξέρουμε ότι το πακέτο για την καθαρή ενέργεια αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμα νομοθετικά προσκόμματα που πρέπει να αρθούν. για την εξομάλυση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την ενεργειακή αποθήκευση και φυσικά έχουμε και την ασφάλεια φωδιασμού που πάντα μας απασχολεί. Για τις μπαταρίες ξέρουμε ότι κατέχει το 50% των ε, ε, επιχειρήσεων ε, εξόριξης λιθίου και κοβαλτίου. Υπάρχει μετά και το ζήτημα της, των εθνικών μέτρων στήριξης σε σχέση με την ανάπτυξη των ε, υποδομών και καταστάσεων αποθήκευσης και να δούμε τι πρέπει να αλλάξει ε, στο επόμενο καθεστώς ε, για τις κρατικές ενισχύσεις την περίοδο μετά το 2022. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, σκιώδης από την ΚΟΕ, ο κύριος Γεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη διαλεκτική της στάση και διάθεση να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος το οποίο θα μπορούσε να επουλώσει κάποιες από τις πληγές της κλιματικής αλλαγής. Ο πλανήτης μας έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά και ό,τι δεν κάηκε ακόμη χάνεται στις πλημμύρες. Για να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει απαιτούνται δραστικά μέτρα επιτέλου. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποθήκευση ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για επίδευξη ενό ενεργειακού συστήματο με μηδενικέ εκπομπέ, το οποίο να βασίζεται αποκλειστικά στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Έχουμε ακούσει βαρύκλουπε εξαγγελίε, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε απαιτούνται μέτρα, όχι άλλα λόγια και υποσχέσει. Η ενέργεια είναι έναν αναντικατάστατο κοινωνικό αγαθών και πρωταρχικό στόχο θα πρέπει να είναι η αποθήκευση ενέργεια να λειτουργήσει ω ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια και καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια. Είναι επίση αδύρυτη ανάγκη να διασφαλίσουμε πω όλοι οι πολίτε θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και δυνατότητα να αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποθήκευση ενέργεια. ιδιαίτερη στήριξη πρέπει να δοθεί κατά την άποψή μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών αποθήκευση. Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω μεταβατικό καύσιμο, το τονίζω, ω μεταβατικό καύσιμο μέχρι την επίτευξη του στόχου για πλήρη στροφή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Προ αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και οι τροπολογίε που θα καταθέσουμε ενό πολιτική ομάδα σε συνεργασία με την εισηγήτρια αλλά και με του συναδέλφου σκιώδη εισηγητέ. Είμαι βέβαιο ότι θα εργαστούμε παραγωγικά και θα πετύχουμε συλλογικά το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέσσερις ε, παρεμβάσεις ε, του ενός λεπτού από τους συναδέλφους, πέντε. Τρία λεπτά στο τέλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια θα δώσουμε το λόγο και στην εισηγήτρια, στην κυρία Γαμών. Πεκαρίνεν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ζητήματα. Συσσωρευτές ε, και CCS. Α, βασιζόμαστε πάρα πολύ στην παραγωγή από την Κίνα. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας. Πάνω από το 60% της παραγωγής κοβαλτίου προέρχεται λοιπόν από την ε, Κίνα, που είναι πολύ σημαντικό υλικό για, την, ε, για το θέμα που μας απασχολεί. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο δράση που είναι το πρώτο βήμα διόρθωσης των ενεργειών μας, όμως χρειαζόμαστε ε, περισσότερες ενέργειες από αυτή την άποψη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει περισσότερο δράση από ό,τι τώρα. Και μετά για την ε, ε, δέσμευση και αποθήκευση θεωρούς, ανθρακά, θεωρούσαμε πριν από 10-15 χρόνια ότι θα αποτελούσε την απάντηση στα προβλήματά μας, όμως αυτό δεν συνέβη. Τώρα που οι τιμές του τόνου διοξιδίου του άνθρακα είναι 25-30 ευρώ τον τόνο, βλέπω ότι μπορεί σε μερικά χρόνια να δημιουργήσουμε αυτές τις τεχνολογίες ε, CCS. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε, μάλλον κατά την ε, κατάρτιση του προγράμματος Horizon, να διατηρήσουμε κάποια κονδύλια για αυτό το ζήτημα, ελπίζω σε μερικέ δεκαετίες να είναι περιττό, να μην χρειαζόμαστε αυτή την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα. Αλλά για τα επόμενα 20-30 χρόνια ίσως θα πρέπει να χρειαστεί να αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία. Σε αυτή την ε, έκθεση της πρωτοβουλίας καλό είναι να βρούμε νέες ε, ιδέες, να τις προωθήσουμε και στην Επιτροπή μας και μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Έξι συνάδελφοι μάλλον έχουν στήσει το λόγο. Κουπλανάτρι τώρα. Ευχαριστώ. Γίνεται μια καλή έκθεση πρωτοβουλίας με μεγάλο εύρος. Η δυσκολία είναι κάπως να περιορίσουμε το πεδίο. Ξέρουμε πολλά για τους ε, συσσωρευτές. Ε, ο Σεύκοβιτς ακόμα ε, είναι αρμόδιος για την προώθηση της πολιτική για τι ενώσιμε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα. Έχουμε ανθρακοριχεία ε, που δεν ε, ε, χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούμε ακόμα ορυχία, μάλλον, όχι και χρησιμοποιούμε ακόμα άλλα από την Αφρική. Το ίδιο ισχύει και με πρώτες ύλε που έρχονται από την Ασία να θα μπορούσαμε να έχουμε από εδώ. Χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα από το ρηχείο μέχρι την ανακύκλωση και θέλουμε και αυτά τα ανακυκλωμένα ε, υλικά να γίνουν νέα πρώτη ύλη. Αυτή η έκθεση μπορεί να κάνει τη διαφορά σε σχέση με την άσκηση της πίεσης για τη μεταρρύθμιση, αναθεώρηση του κανονισμού για ε, τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ε, σε ό,τι έχει να κάνει με ε, τους ισορρευτές, ε, την αποθήκευση και την θέρμανση και ψήξη. Μετά έχουμε να κάνουμε και με τις πρώτες ύλες. Κάποιες φορές σκεφτόμαστε μόνο την θέρμανση ύδατος, αλλά υπάρχουν... Εγώ μιλώ με άλλους επιστήμονες που βρίσκουν και άλλους τρόπους πέρα από το νερό. Ευχαριστώ, κύριος Μπούκνερ από τους Πράσινους. Vielen Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ στην αποθήκευση μεγάλων ογκών ενέργεια, στη σταθεροποίηση του δικτύου και ε, στις ανάγκες της βιομηχανία. Εδώ, λόγω της ε, δυνατότητας αποθήκευση και της πυκνότητας ενέργειας, έχουμε περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευση. Ε, πολλές φορές ακούσαμε το υδρογόνο ως πηγή αποθήκες, ως πηγή ενέργειας. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης δεν παράγεται μόνο υδρογόνο, αλλά και διάφορες ε, άλλες ουσίες. Έπειτα, ε, μια δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι θα πρέπει να εργαστούμε διατομεακά. Η ηλεκτροληση σε υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί, ε, αποθήκευση, δημιουργεί παραγωγή ρεύματος ε, που είναι κατά 60%, μας γυρίζει κατά 60% πίσω. Ανακτάται δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η μέθοδος όμως λειτουργεί μόνο όταν συνδυάζεται με διάφορες άλλες, με την, με την χρήση του υδρογόνου ας πούμε στην ε, χαλιβουργία. Ε, Γι' αυτό λοιπόν, με λίγα λόγια, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση να εξεταστεί το θέμα διατομεακά και όχι μεμονωμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούχνερ. Ο κύριος ε, Κοφούτ, εκ μέρου των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες και να τους δείξουμε κατά πόσον είναι αποτελεσματικά όλα αυτά τα προγράμματα. Στη Σιλεσία πάντα είχαμε κοινωνική διαβούλευση. Η κυβέρνηση μάλιστα αποφάσιζε ποιον θα επιδοτούσε και όχι. Αυτά τα πράσινα project στην Ευρώπη θα μπορούσαν επίσης να υποβληθούν σε διαδικασίες διαβούλευσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν συνέχεια να πληρώνουν την ύφη για τα project, παρά μόνο σε περίπτωση που δώσουν την άποψή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκα, ε, συγγνώμη που δεν σας είδα νωρίτερα. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσω τη γλώσσα μου. Θα μιλήσω ορμανικά. Θέλω να μιλήσω για την αποθήκευση ενέργειας. Μέχρι στιγμής ε, αυτό το θέμα ε, θεωρούνταν ταμπού. Χρειάζεται μια επαρκής τεχνολογία, μια τεχνολογία αποθήκευσης ε, επαρκής. Έχουμε την ε, Πράσινη Συμφωνία, έχουμε την, τους στόχους απομάκρυνσης από το διοξίδιο του άνθρακα, χωρίς την αποθήκευση, δυνατότητα αποθήκευση, δεν μπορούμε σοβαρά να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Μέχρι στιγμή το 1% μόνο τη ισόρρευση δεν είναι υδροηλεκτρικό. Έχουμε 180 χρόνια ε, υδροηλεκτρικής ενέργειας και την αποθηκεύουμε. Εντάξει. Αλλά θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ε, πηγές ενέργειας ε, από τις οποίες αποθηκεύουμε και θα πρέπει να τι αναπτύξουμε σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση, θα πρέπει να υπάρχουν φορεί που θα ασχολούνται με την αποθήκευση τη ενέργεια. και θα πρέπει να είναι φορεί στον τομέα τη Ευρώπη της, ε, της ενέργειας. Το ορίζοντα Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει μαζικά σε αυτέ τι ε, προηγμένες τεχνολογίε, γιατί θα μπορούσαν να μας δώσουν πραγματικές λύσεις ε, για την αποθήκευση. Έχουμε τις ηλεκτρικές μπαταρίες αλλά δεν είναι οι ηλεκτρικέ συστοιχίε, αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Μιλήσαμε για το υδρογόνο, έτσι. Στα πλαίσια της νέας πράσινη συμφωνία, το υδρογόνο θα είναι μία από τις πιο σημαντικές λύσεις. Ε, θα υπάρχουν και άλλες λύσεις, αλλά δεν είναι ακόμα πολύ παρούσες στη ζωή μας, γιατί θεωρούνται πολύ ακριβές. Ακριβές τι σημαίνει. Ότι υπάρχει δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουμε, απλώς πρέπει να χαμηλώσουμε την τιμή. Ε, ο συντονιστής ε, του ΕΛΚ. Ήδη ακούστηκαν πολλά για, τις, για τα προτερήματα και τα μενεκτήματα της τεχνολογίας αυτής. Το δύσκολο είναι ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε μεμονωμένα τις τεχνολογίες αποθήκευσης, αλλά να εξετάσουμε και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Όπως ακούσαμε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να τις εξετάσουμε ως κομμάτι της βιομηχανικής στρατηγικής. Ίσως ε, Λοιπόν, μιλάμε πάντα για τεχνολογία, όμως ε, βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη δεν είναι η ίδια η προθυμία όλων ε, και δεν υπάρχει πάντα το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας. Υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια με τον ε, παραδοσιακό ε, τρόπο, υπάρχουν άλλες που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους. Θεωρώ πάντως πως σημαντικά είναι τα εξής. Όταν καταρτίζουμε μία βιομηχανική στρατηγική πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε όλες τις απόψεις. Δεν έχει νόημα λοιπόν να χρησιμοποιούμε το power to gas ενέργεια σε αέριο χωρίς να συνυπολογίζουμε και την χρήση του στις ε, μεταφορές. Ε, οι μεταφορές ε, χαρακτηρίζονται από κινητικότητα. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς, να δούμε το σύνολο της αλυσίδας αξίας και να αναγνωρίσουμε ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η αντίσταση των κρατών μελών στην αποθήκευση ενέργειας. Πολύ ωραίες οι τεχνολογίες και οι καινοτομίες, όμως αν δεν υπάρχει το πλαίσιο δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασάρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι τόσο η συγγήτρια όπως και οι υπόλοιποι, ε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για να προχωρήσουμε στην ε, απανθρακοποίηση, στην απεξάρτηση από το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ανανεώσιμη ενέργεια έχουμε. Έχουμε δύο δυνατότητε ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καταρχάς πρέπει να έχουμε καλές διασυνδέσεις. Έτσι. Τι έχουμε στη Γαλλική, ας πούμε, στην Ισπανία κτλ. Ε, που δεν έχουμε αρκετό ήλιο, ε, θα πρέπει να συνδεθούμε με περιοχές της Ισπανίας, ας πούμε, που έχουν πολύ ήλιο. Άρα, καλές διασυνδέσεις είναι το πρώτο. Και δεύτερον, αποθήκευση. Πολύ σημαντικό. Κάνω μια έκκληση να ξεκινήσουμε με την ε, ηλιακή ενέργεια. Πολλές ε, χώρες έχουμε ηλιακή ενέργεια, μειώθηκαν οι τιμές και πουλάμε και την ε, ηλιακή μας ενέργεια, θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε τις, ε, τις χώρες να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές για να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις τεχνολογίες και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες. Θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Από το Renew, Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται εκφύσεως και πολλέ τεχνικέ δεν είναι όριμε για να φτάσουμε ε, σε λύσεις ε, αποθήκευσης. Ε, άρα θέλουμε καινοτομία. Άρα θα πρέπει να διερευνήσουμε όλε τι δυνατότητε που έχουμε και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια μια ευρωπαϊκή συμμαχία. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο και τη στρατηγική, νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε Πρέπει να δούμε μαζί με το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν ε, τις ε, ευρωπαϊκές συμμαχίες, όπως παραδείγματος χάρη στην, ε, στην μπαταρία, στις μπαταρίες, καινοτομίες που δεν θα χρησιμοποιούν, ας πούμε, ούτε λίθιο ούτε κοβάλτιο Η Κομισιόν θα μας μιλήσει για μια νέα ευρωπαϊκή συμμαχία για το υδρογόνο είναι ακόμα ένα θέμα που οι διάφορες χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να φτιάξουν ένα κλάδο ε, που είναι στα σπάργανα. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στο Στρασβούργο όλοι ε, και χάσαμε την ειδική μερίδα που έγινε για αυτό το θέμα. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε το δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας στο διάστημα. Σας φαίνεται βλακώδες, αλλά το διάστημα είναι θαυμάσιο για τις ε, ηλιακές στοιχείες. Ε, θα μπορούσαμε ας πούμε, να βρούμε λύση εκεί πάνω, στο διάστημα, όπως προτείνουν οι Κινέζοι. Θα μπορούσαμε να παράγουμε και να ε, δαπανάμε πολλή ενέργεια. Παραδείγματο χάρη τα data center, τα οποία εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όλη την αεροπορία του κόσμου, του πλανήτη. Έτσι. Αλλά όμως η, εκπομπή αυτή του διοξιδίου του άνθρακα στο, στο διάστημα γίνεται πολύ πολύ μακριά. Και επίσης ε, μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ηλιακές στοιχείες εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεφτά τη συζήτηση για το διάστημα. Θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια και εκεί. Θα ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Στέφαν Μότζερ από την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΝΕΡ ε, τμήματάρχης για την ενεργειακή ασφάλεια. Τρία λεφτά μάγιστο, μέγιστο διάστημα. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ, εκ μέρου τη Επιτροπή. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση ιδία πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για την αποθήκευση ενέργεια, για να δοθεί πολιτική καθοδήγηση για το πώ θα προχωρήσουμε, τι πρέπει να μα απασχολήσει και σε τι να επικεντρωθούμε και πώ θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Το πακέτο καθαρή ενέργεια είναι η βάση, πολλά έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα θα πρέπει να το δούμε στο τμήμα της προσπάθειας για την Πράσινη Συμφωνία, όλη η Ένωση να κάνει περισσότερη προσπάθεια για να είναι πιο φιλόδοξη και το, η αποθήκευση ενέργειας είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίσει ε, ασφάλεια νεφοδιασμού, όπως ανέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτές. Πρέπει να δούμε τι άποψη έχει η αγορά με βάση τις ανάγκες αγοράς, αλλά χρειάζεται στήριξη αγορά από ένα πολύ καλό και επαρκέ ε, κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη που παίζουν κρίσιμο ρόλο ε, στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων κλίματος και ενέργειας για να βελτιώσουν τους κανόνες για, για την αποθήκευση, πόση αποθήκευση χρειάζεται, ε, με βάση την εθνική, τις εθνικές ιδιαιτερότητες όπως ανέφεραν και πολλοί ευρωβουλευτές. Δεν είναι η ίδια κατάσταση εξάλλου σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορετικές αδυναμίες και ισχυρά σημεία γεωγραφικά ε, διάθεσης ε, ενεργειακών ε, πόρων κτλ. Και ίσως θα πρέπει να δώσουν και εθνική στήριξη. Γιατί έχουμε ευρωπαϊκή στήριξη από τον ορίζοντα 2020, τον ορίζοντα Ευρώπη, αλλά και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας για project έργα δηλαδή υποδομών, αλλά ίσως θα χρειαστούν και εθνικά, εθνική στήριξη. Θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για να κατευθύνουμε Καλύτερα το τι πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, όπως αναφέρθηκαν, ανέφεραν και οι βουλευτές. Τώρα δεν είναι δυνατόν να επιλέξουμε την καλύτερη τεχνολογία. Χρειαζόμαστε στρατηγική προσέγγιση, να δούμε τα εμπόδια και να επιτρέψουμε σε όλους τους φορείς της αγοράς, τους πολίτες, επίσης να προχωρήσουν και να επιλέξουν την καλύτερη λύση με βάση τις διαφορετικές ανάγκες που έχουμε. Όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να υπάρχει και στενή συνεργασία παντού, διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μοιραστούμε τους πόρους μας, θα πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση επάρκειας για να δούμε αν υπάρχει ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασμού, πού πρέπει να αποθηκεύεται η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να εξασφαλίσουν την συνολική ασφάλεια του συστήματος σε ηλεκτρική ενέργεια, προχωρώντας προς ένα σύστημα που δεν θα έχει καθόλου εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ, θέλω να συνεργαστούμε. Η Κομισιόν κάνει και μια μελέτη με εξωτερικούς συμβούλους, με σκοπό να φτάσουμε σε κάποιες συστάσεις, τις οποίες θα ενσωματώσουμε στη στρατηγική για έναν έξυπνο τομέα ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Μόζερ. Η συγγήτρια θα απαντήσει τώρα και θα φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους και τις απόψεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μόζερ για τα σχόλιά του. Ελπίζω τα αποτελέσματα της μελέτης να συμπεριληφθούν στην έκθεση, διότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνολική εικόνα για τις δυνατότητες αποθήκευσης που διαθέτει η κάθε χώρα. Θα σχολιάσω κάποια λίγα πράγματα για να μείνω εντός χρονικού ορίου και θα γυρίσω στη γλώσσα μου. Κύριε Έλερ, λοιπόν, δεν ε, πρόκειται για απαρίθμηση των τεχνολογιών αποθήκευσης. Δεν ήθελα να κάνω αυτό. Ήθελα όμως να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες. Υπάρχει αγορά, όπως αναφέρατε κι εσείς. Και σε ορισμένα σημεία που συμφωνώ μαζί σας ε, και στην Αυστρία είναι πολύ συχνά ε, δύσκολο να ε, προχωρήσουμε τεχνολογικά διότι πάντα θα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Η πολιτική βούληση είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι πολιτικοί έχουν καθήκον να ενημερώνουν τους πολίτες και σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχουν άλλα πολύ καλά παραδείγματα με την, ε, όπου η πολιτική ενημερώνει τους πολίτες. Ε, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, αλλά στην Ελβετία έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έχει συνεργαστεί η πολιτική με τους πολίτες ε, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην πρόοδο ενωμένοι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ευθύνη των πολιτικών. και μάλιστα οι αντλίες ε, αποθήκευσης είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές σαν τεχνολογία. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν έχουμε μια σχεδόν πολυτέλεια να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, γιατί δεν το κάνουμε. Ας μην ε, κοιτάμε μόνο λοιπόν τα θετικά παραδείγματα, αλλά ας δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και να την προσαρμόσουμε στην ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να βρούμε μια καλή λύση και να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα των διαθέσιμων τεχνολογιών. Είναι μια πρόκληση, σίγουρα αυτό, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, αλλά θεωρώ πως η πρόταση να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθεί η αποθήκευση ενέργειας με την βιομηχανική στρατηγική είναι πάρα πολύ καλή σίγουρα θα έχει η βιομηχανία να μας δώσει πολλά. Κύριε Πούχνερ, δεν περιοριζόμαστε μόνο στο υδρογόνο. Αυτό δεν θα ήταν συνετό έτσι κι αλλιώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνεργαστούν όλοι οι τομείς, να είναι διατομιακή αυτή η προσπάθεια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα αποτελέσει πολύ σημαντικό κομμάτι του όλου εγχειρήματο. Και για να ολοκληρώσω στις ε, γερμανικές ε, απαντήσεις, θα ήθελα να πω στην συνάδελφο ότι καταλαβαίνω πως η ενεργειακή ασφάλεια, η ασφάλεια εφοδιασμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν το αρνούμε και εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να παρέχουμε αυτή την ασφάλεια. Όμως ε, νομίζω πως ε, αυτό συνδέεται άρρηκτα με την αποθήκευση της ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς ε, όπου στερούνται δοτικότητας, όπου δεν και γι' αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μορφές θέρμανσης όπως τις αντιλές θερμότητας ή τη τηλεθέρμανση όπως κάνουμε ήδη στη Γερμανία. Και συνεχίζω στα αγγλικά. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους, όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές και τους ε, εξαιρετικούς βοηθούς και εμπειρογνώμονες στην ε, συνάντηση που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες Είχατε πάρα πολλά να συνεισφέρετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι το εγχείρημα αυτό. Η ενεργειακή μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική για να είμαστε διχασμένοι. Δεν θα μακρηγορήσω για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Θα πω όμω ότι η πρώτη μας συνάντηση ήταν επικοδομητική και ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, δουλειά σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας. Σήμερα είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα περάσουμε από την αποθήκευση ενέργειας στο διάστημα ένα κομμάτι της ε, όλης άσκησης της ε, Επιτροπής μας είναι να καλέσουμε τους ε, διάφορους οργανισμούς που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για συζήτηση. Καλωσορίζω λοιπόν τον Καλός Λεωρίδες από τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS Και να πω ότι η αρχική μας πρόθεση ήταν να είχαμε και τους διοργανισμούς ε, του και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά ο κύριος Βέρνερ, Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Συμφωνήσαμε όμως ε, να τον καλέσουμε σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας, το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Όμως ο κύριος Τεσορίδας είναι παρόν και προτείνω, μια που έχουμε εκπρόσωπο μίας ε, όμως ε, υπηρεσίες ενός οργανισμού να περιοριστούμε στην ε, μία ώρα, διότι στις μία και μισή θα έρθει η Επίτροπος Βεστάρ και θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει να μας πει. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα να το κάνουν ήσυχα. Κύριε Τεσορίδες, είστε ο ευθύς του Ευρωπαϊκού GNSS, του GSA. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο, αλλά πριν θα ήθελα να πω ότι δεν θα συζητήσουμε το θέμα του Γκαλιλαίου σήμερα, διότι εκεί ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Το ζήτημα αυτό θα το εξετάσουμε ξεχωριστά σε δεύτερο χρόνο, κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Φεβρουαρίου. Προτείνω λοιπόν να εργαστούμε ω εξή. Ε, να ξεκινήσει ο κ. με μια παρέμβαση 10 λεπτών, να μα εξηγήσει ε, τι προτεραιότητε του οργανισμού του, τις ε, προκλήσει και να μα εκθέσει τα απόψει του για τα κύρια θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια να καλέσουμε τους συντονιστές τους ε, αντικαταστάτες τους και έπειτα όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να υποβάλουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια. Στη συνέχεια ο κύριος Δεστορίδας θα απαντήσει και θα κάνει τα κατακλητικά του σχόλια. Αν έχουμε χρόνο, μια που είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον θέλει να μιλήσει, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μετά θα ζητήσω ε, σε όποιον από εσάς το επιθυμεί να δευτερολογήσει. Κύριε Τελωρίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε σήμερα και σας δίνω το λόγο να, για να μας παρουσιάσετε τις δραστηριότητες του οργανισμού σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σας μιλήσω εξ ονόματος ε, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, αλλά και του Οργανισμού και του Παγκοσμίου Διορφορικού Σύστημα Πλοήγησης. Σε αυτή τη δεκάλεπτη εισήγηση θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για τον οργανισμό μας ε, και τα επιτεύγματά του. Μετά, να, θα ήθελα να σταθώ στα όσα προκύπτουν από τον κανονισμό που θα τεθεί σε ισχύ από τον ε, επόμενο Ιανουάριο. Τα νεότερα δηλαδή για τους ε, δύο οργανισμούς και τέλος να σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της αγοράς. πώς έχει η κατάσταση και τι προβλέπετε για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, για τον GSA είναι ένας οργανισμός λοιπόν που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία 8-9 χρόνια. Έχουμε περίπου 200 μέλη του προσωπικού. Όχι μόνο στην έδρα μας, στην Πράγα, εκεί βέβαια είναι η πλειονότητά τους. Έχουμε όμως και επιχειρησιακά κέντρα κοντά στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στις κάτω χώρες και ένα γραφείο στην Τουλούζ. Δύο επιχειρησιακά κέντρα ασχολούνται συγκεκριμένα με την ε, παρακολούθηση της ασφάλειας του συστήματος. Και επισημαίνω εδώ ότι στελεχώνονται από το προσωπικό μας επί 24 ώρου βάσεως. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τους δύο βασικούς πυλώνες του οργανισμού μας. Πρώτα έχουμε την παροχή υπηρεσιών. Για το έγνος, που είναι ένα περιφερειακό σύστημα που αφαιρά την Ευρώπη και αυξάνει την απόδοση του GPS κυρίως για την πολιτική αεροπορία και παροχή υπηρεσιών για τον Γαλιλαίο. Αναλάβαμε αυτή την αρμοδιότητα από την 1η Πρώτου 2017 και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ανάληψης αυτής της αρμοδιότητας ε, είναι να σας μιλήσω για την ε, παρίσπιση στην αγορά. Το έγνος από το 2011 που τέθηκε σε ισχύ σε 9 χρόνια περίπου. Βλέπουμε ότι σήμερα έχει το 50% των ε, επιχειρησιακών αεροδιαδρόμων στην Ευρώπη. Και όλες οι μεγάλες εταιρείες ε, κατασκευής αεροσκαφών, όπως η Airbus και η Boeing, προσφέρουν ε, νέα αεροσκάφη με το σύστημά μας, με το έγνος. Πάνω από 350 αεροδρόμια λοιπόν σε όλη την Ευρώπη ωφελούνται αυτής της, επωφελούνται από αυτή τη νέα τεχνολογία. Θεωρείται μεγάλη τομή ε, στην τεχνολογία, μεγαλύτερη μετά από την εφεύρεση του ραντάρ. Τώρα, για το πρόγραμμα Γαλιλαίος. ήταν μια νέα αρμοδιότητα που ανέλαβε ο οργανισμός υπό την παροχή υπηρεσιών προς τον Γαλιλαίο. Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε φτάσει τα ένα δις συσκευών, κυρίως smartphone, που είναι ε, συμβατές με το Γαλιλαίο. Είναι λοιπόν μια τεράστια επιτυχία τον Γαλιλαίο τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα υπερβαίνουν και τις ε, προσδοκίες μας πριν από 3-4 χρόνια. Πού οφείλεται αυτή η επιτυχία? Σίγουρα ένα ε, σύστημα που λειτουργεί αρκετά καλά, προσφέρει κάτι επιπλέον κάτι καινούριο σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα πλοήγησης ανά τον κόσμο και σίγουρα η επιτυχία οφείλεται σε έναν βαθμό και στις ενέργειες του οργανισμού. Δεν φτάνει μόνο να αποστέλουμε ένα μήνυμα στο διάστημα, το κύριο είναι πώς θα φέρουμε το μήνυμα σε επαφή με τον ε, χρήστη. Αυτό είναι ο βασικός παράγοντας για την πρόσληψη στην αγορά. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν στους ε, χρήστες, να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους, να τους βοηθήσουμε να ε, πάρουν μια απόφαση. Σας μίλησα για το ένα δις συσκευών. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μια τεράστια επένδυση και από τους ε, κατασκευαστές microchip, και εκεί υπάρχει το ζήτημα του γιατί επέλεξαν τον Γαλιλαίο. Οι επιχειρήσεις αυτές λοιπόν θεώρησαν ότι ο Γαλιλαίος τους προσφέρει δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική στην αγορά. Τους προσεγγίσαμε λοιπόν, κατανοήσαμε τις ανάγκες τους και εκείνοι δοκιμάζουν τις συσκευές και από οικονομικής άποψης, όποτε αυτό είναι δυνατόν, τους βοηθούμε να μπουν στην αγορά. Το καλύτερο στοιχείο που μπορώ να σας δώσω είναι το εξή. Μπορεί να γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο περίπου ο οργανισμός εκδίδει μία έκθεση αγοράς. Η οποία γρήγορα γίνεται σημείο αναφορά σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορείτε να το βρείτε και στον ιστότοπο του οργανισμού GSA, δωρεάν φυσικά. Θα σας δώσω λοιπόν μια εικόνα Τις πρώτες 100 ημέρες της δημοσίευσης της έκθεσης έχουμε, έχουμε μάλλον περίπου 10.000 downloads σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν ε, ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τη γνώση που έχει να παρέχει ο GSA. Ολοκληρώνοντας το κομμάτι αυτό θα ήθελα να μιλήσω για την διάσταση της ασφάλειας, που είναι επίσης σημαντική για το πρόγραμμα GNSS. Όχι μόνο επειδή ένα από τα, από σήματα είναι κρυπτογραφημένο, που αφορά μόνο ε, τους θεσμικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένης και της άμυνας, αλλά όλο ένα και περισσότερο η ασφάλεια παίρνει μεγαλύτερη σημασία πια για οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα. Ε, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα μελήματα, αλλά για ένα σύστημα που έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι θεμελιώδες. Για να καταλάβετε, η πρόσφατη ανάλυση μας δείχνει ότι περίπου 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ συνδέεται με κάποιον τρόπο με το GNSS. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ο κανονισμός. που θα τεθεί σε ισχύ σε περίπου ένα χρόνο. Που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα συνολικό ε, νομικό πλαίσιο. Να σας πω εν συντομία γιατί είναι τόσο σημαντικό για τον οργανισμό μας. Πρώτον, γιατί αξιοποιεί την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια προ όφελο άλλων προγραμμάτων. Πρώτα απ' όλα, ο GSA αφήνει κατά μέρο ε, την εστίαση στην πλοήγηση και γίνεται νέος ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Διαστημικού Προγράμματος, όπως και άλλα προγράμματα, όπως ο Κοπέρνικος, το GovSatcom, SSA. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρώπη ωφελείται από την εμπειρία που έχει αποκομίσει ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της ασφάλειας και στα αποτελέσματα στην αγορά. Φυσικά με τα χαράς θα επανέλθω. Τώρα, για τα αποτελέσματα στην αγορά. Είχαμε αρχικά τεράστια αγορά των ε, smartphone. Πάνω από 30 εταιρείες προσφέρουν συμβατότητα με το Γαλιλαίο. Γίνεται σταδιακά de facto μάλιστα το στάνταρ σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε 25 μάρκες αυτοκινήτου που στα νέα τους μοντέλα θα έχουν το Γαλιλαίο. Αυτό συνάδει και με, την, ε, το σχετικό κανονισμό που τέθησε ισχύ τον Απρίλιο 2018, αλλά μιλώ και για όλα τα μελλοντικά αυτόνομα αυτοκίνητα, όλες ε, οι μεγάλες ε, εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας δοκιμάζουν το Γαλιλαίο. Πριν από μερικές εβδομάδες στην Κομπιάνγκ δοκιμάσαμε ένα αυτόνομο ε, όχημα με επίπεδο αυτοματοποίησης σε 4 από τα 4 στα 5. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας για το Γαλιλαίο και το έγνος. Στην αεροπλοεία, ήδη σας είπα ότι πρόκειται για τομή στην τεχνολογία. Ε, στα μη επανδρομένη αεροσκάφη, που είναι ένας ραγδαία πτυσσόμενος τομέας, ήδη έχουμε πάνω από 150 μοντέλα από 35 κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το έγνωση του Γαλιλαίου. Στους σιδηροδρόμους, Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 40.000 βαγόνια με χρήση του Γαλιλαίου για την ε, διαχείριση στοιχείων. Η πρόκληση βεβαίως εδώ είναι η χρήση του Γαλιλαίου και το έγνος ε, για την αποστολή σημάτων στους σιδηροδρόμους. γιατί στους σιδηροδρόμους δεν έχουμε μεγάλη τάση προς την καινοτομία. Υπάρχει κάτι κερματισμός, είναι δύσκολο να ε, παρακάμψουμε αυτά τα εμπόδια. Για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, 20% των υποδοχέων, των δεκτών μάλλον, ε, χρησιμοποιούν τον Γαλιλαίο. Ε, θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να σας έχω δώσει μια εικόνα της επιτυχίας ε, του Έγνους και του Γαλιλαίου μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεσδορίδες. Πολύ σαφή, συνοπτική και ενημερωτική αυτή η παρουσίαση με ενδιαφέροντα στοιχεία και παραδείγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Το λόγο τώρα θα λάβουν ε, τα μέλη μας ε, για σχόλια, ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ξεκινούμε πάντα από τους συντονιστές. Φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και η γραμματεία θα σημειώσει τα όνοματά σας. Από τους συντονιστές ο κύριος Σάιλερ πρώτος. Ο κύριος Σαλίνη θα πάρει το λόγο εξ ονοματάζους μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Σαλίνη είναι εισηγητής για το διαστημικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεστορίδε. γιατί κλείνει ως διευθυντής ε, για το GSA, ε, στο GSA. Κλείνει τη θητεία του, τελειώνει τη θητεία του. Έχουμε πολλές προκλήσεις, τώρα μιλάμε όμως για τον προϋπολογισμό. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω από τα λεφτά. Ξέρουμε ότι είπα αποφάσισαν να επενδύσουν 22,6 δισεκατομμύρια ε, δολάρια μόνο για το 2020 για το διάστημα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την πρότασή μας 16 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί χωρίς επενδύσεις δεν μπορούμε να μιλάμε για το διάστημα στο μέλλον στην Ευρώπη η, απόφαση του ESA τη Υπηρεσίας Διαστήματος, για ένα προπολογισμό 14,5 δισεκατομμύρια για τρία χρόνια είναι, μια... είναι καλέ ειδήσει, καλά νέα για μα, αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση, ω GSA ή e USPA στο μέλλον, να έχουμε ένα καλό προπολογισμό για να επενδύσουμε και για να διατηρήσουμε τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο ως παλιά και παραδοσιακά προγράμματα και να επενδύσουμε για νέα, σε νέα προγράμματα, το COFSATCOM και τα λοιπά. Για να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να μιλάμε με μία φωνή ως Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες χώρες έχει προσέγγιση που εστιάζει στην άμυνα, ενώ άλλες χώρες έχει μια προσέγγιση μη στρατιωτική. Αλλά έγινε και ε, συζήτηση στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία για τη διαχείριση, για τη διακυβέρνηση και προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε κοινή προσέγγιση. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο τελευταίο τμήμα των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό και να κλείσουμε και τις συζητήσεις για την διακυβέρνηση. Γιατί Ακόμα έχουμε πολλές αγγίλες ανοιχτέ που δεν τι έχουμε κλείσει, πολλά σημεία που δεν έχουμε κλείσει. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξο. Γιατί εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε καλή γενική προσέγγιση για το διάστημα, για αυτά τα προβλήματα. Δεύτερον, που είναι η, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το διάστημα. Κατά την άποψή μου είναι αρμοδιότητα στη ΣΥΤΡΕ. Ε, και το βασικό μας θέμα είναι η βιομηχανία. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους πολίτες και μπορούμε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ε, εξατομικευμένα στους πολίτες μας. Είναι κρίμα, γιατί συχνά οι πολίτες μας θεωρούν ότι το GPS είναι μια υπηρεσία που παρέχει ο Γκαλιλαίο. Πρέπει να επενδύσουμε για τους πολίτες μας. Πρέπει να επενδύσουμε σε επικοινωνίες. Οι επικοινωνίες δεν είναι ένας τρόπος να πληροφορούμαστε μόνο. Είναι στοιχείο της πραγματικής δημοκρατίας. Είναι γεωπολιτικά σημαντικό, γιατί αν οι πολίτες, ας πούμε, δεν γνωρίζουν ότι επενδύω για αυτούς, πώς θα επιλέξουν την Ευρώπη, πώς θα είναι υπέρ της Ευρώπης όταν ψηφίζουν, ας πούμε. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις ανάμεσα σε προγράμματα του διαστήματος και άλλα σημαντικά προγράμματα, όπως α πούμε την Πράσινη Συμφωνία. Ένα πρόγραμμα για το διάστημα είναι σημαντικό για να έχουμε καλά αποτελέσματα στην Πράσινη Συμφωνία. Ο Κοπέρνικος έχει πολλά εργαλεία <coughs> για να βελτιώσει την Πράσινη Συμφωνία. Για, την για το ψηφιακό θεματολόγιο επίσης. Χωρί τα αποτελέσματα του προγράμματο για το διάστημα, υπάρχει κίνδυνο η πράσινη συμφωνία ή το ψηφιακό θεματολόγιο να παραμείνουν απλά σλόγγαν, γράμματα κενά περιεχομένου. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αλληλοσύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά διαφορετικά προγράμματα. Και επίσης χρειαζόμαστε και διεθνή συνεργασία. Την τελευταία περίοδο Στον ορίζοντα Ευρώπη, συγγνώμη, στον ορίζοντα 2020 διορθώνει ο είχαμε μία ειδική γραμμή για το διάστημα. Τώρα, στον ορίζοντα Ευρώπη, δεν έχουμε ειδική γραμμή προϋπολογισμού για το διάστημα. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί όταν είσαι επενδυτή από μια τρίτη χώρα ξέρει ότι έχουμε νομικό και ρυθμιστικό ξεκάθαρο πλαίσιο για το διάστημα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει την επένδυση. Και ο Ευρωπαίος επενδυτής και ο ξένος επενδυτής. Το ίδιο ισχύει και για τους δύο. Άρα θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε και αυτά τα θέματα και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλές προκλήσεις. Ε, εμείς θέλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κλείσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουμε με μια νέα πραγματική πρόταση για το διάστημα και να δημιουργήσουμε καλή σχέση, κατά την άποψή μου, ανάμεσα στα προγράμματα για το διάστημα και τα προγράμματα για την άμυνα. Να έχουμε μια προσέγγιση μη στρατιωτική, αλλά να έχουμε καλή σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο προγράμματα, που είναι διαφορετικά, αλλά και συνδεδεμένα και συμπληρωματικά. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλίνη. Ο κύριος Κρούγκερ από Τυρινιού, Ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσει για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Ε, να ευχαριστήσω τον Κάρλο Ντεντορίντε για τι εξηγήσει του καταρχά και να τιμήσω τη δουλειά που έκανε, ε, που κάνει επί πολλά χρόνια στο εσωτερικό της Υπηρεσίας Διαστήματος, γιατί είναι τώρα μια πολύ αναγνωρισμένη υπηρεσία, ένας οργανισμός, πολύ γνωστός, ενώ στην αρχή ήταν άγνωστος. Φτάνετε στο τέλος της θητείας σας, στις 31 Ιανουαρίου, θα παραιτηθείτε από γενικό Διευθυντή, μετά από 9 χρόνια καλών και άξιων υπηρεσιών, το μέγιστο δηλαδή που σας, επιτρέπει, που σας επιτρέπουν οι κανονισμοί. Σήμερα λοιπόν είναι γνωστή η υπηρεσία διαστήματος, η ΕΣΑ. Ε, δύο πράγματα είναι σημαντικά. Ε, δυνατότητες πρόσληψης, είναι περίεργο αυτό, γιατί υπάρχουν δυνατότητες στα διοδρομίας, ε, ποιοτικέ. Και το να προσλαμβάνει η ΕΣΑ ε, προσωπικό ε, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο και είναι κρίμα. Ε, ίσως να έχετε συμβάσεις έτσι αβέβαιες. Ε, ίσως όμως από τις συμβάσεις αυτές θα μπορούσαν κάποιοι να γίνουν έκτακτοι υπάλληλοι. Επίσης υπάρχουν και θέματα προϋπολογισμού εδώ και κάποια χρόνια. Ε, υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπό πρικοδότηση από τη μία τη ΕΣΑ και από την άλλη αύξηση των αρμοδιοτήτων της. Είναι ασύμβατο αυτό. Αν θέλετε να αυξηθεί η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να έχει αυξημένο προϋπολογισμό, ουσιαστικά. Προηγουμένως μιλούσαμε για 200 άτομα που δούλευαν στην ΕΣΑ. στη νέα σας συγγνώμη, ε, που είναι το 10% των, του προσωπικού της ΕΣΑ. Τα θέματα διακυβέρνησης, πρέπει να δούμε. Κάθε ένας έχει ένα ρόλο στις ευρωπαϊκές, ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος. Η Κομισιόν δίνει, έχει το πρόσταγμα, χρηματοδοτεί. Η, ΕΣΑ είναι, κάνει την έρευνα και αναπτύσσει νέα προϊόντα και η υπηρεσία διαστήματος είναι εκεί για το feedback. Θα πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλους τους φορείς. Ε, το διάστημα δεν ε, πρέπει να πέσει θύμα, ας πούμε, πολέμου ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει να τα ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα τα επόμενα χρόνια. Κύριε, ο κ. Σαλίνη μίλησε, μίλησε για τα αυτά τα 16 δισεκατομμύρια προπολογισμού. Εγώ θα είμαι βασιλικότερο του βασιλέου. Θα υπενθυμίσω ότι 16 δισεκατομμύρια είναι η πρόταση τη Κομισιόν, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε 16,9 για το πρόγραμμα διαστήματο. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ψηφίζει τον, τον προπολογισμό, όχι η Κομισιόν, τα 16,9 είναι ο στόχος μας. Έτσι, και εμείς ψηφίζουμε μαζί με το Συμβούλιο. Και με αυτά τα ε, λεφτά μπορούμε να πρικοδοτήσουμε καλύτερα την ε, GSA. Επίσης, από το άρθρο 26 πρέπει να φύγουν ε, οι αγγίλες του, κανονισμού καονισμού δηλαδή του διαστήματος, που μιλάει για την ευρωπαϊκή προτίμηση, για τις, δικέ μας, τις δικές μας βιομηχανίες και εμείς εδώ στην Ιτρέ έχουμε αρμοδιότητες. Πάνω από 50.000 άτομα δουλεύουν στο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλες εταιρείες, σε μικρές εταιρείες, σε μικρομεσαίες και υπάρχει και μια ε, στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα θέματα, κλιματικά, άμυνας, όλα αυτά είναι ένα όλον. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία και ευρωπαϊκή προτίμηση. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο συζήτησε και προτείνει μείον 10% προϋπολογισμό. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα 16,9 δισεκατομμύρια, αλλά και τα 16 καλά είναι. Σας ευχαριστώ που μας τα είπατε όλα αυτά, τα στοιχεία και ευχαριστώ και τον κύριο Σαλίνη. Να κάνω κι εγώ δύο-τρία σχόλια, αν μου επιτρέπετε στο τέλος. Και τώρα πάω στον συντονιστή των Πρασίνων. Κύριε Πέσκα, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά, αλλά γίνεται όλο ένα και σημαντικότερο είναι τα διαστημικά σκουπίδια. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Και από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάποιο πλάνο αντιμετώπισης. Και καθώς μεγαλώνει αυτός ο αριθμός των διαστημικών σκουπιδιών, ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξάνεται αντίστοιχα. Και νομίζω πως ε, θα έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα αυτό που λέτε θα έπρεπε να υπάρχει μία αξιολόγηση κινδύνου έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε και αυτή να περιέχει κάποιες προβλέψεις για το μέλλον, να δούμε αν θα, αυξηθού, θα αυξηθεί ο ρυθμός ή αν θα μειωθεί. Νομίζω πως ε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική απειλή για το διαστημικό πρόγραμμα στο μέλλον και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζωρίνιο για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ για την ε, θαυμάσια δουλειά που κάνει η υπηρεσία διαστήματος. Γιατί χάρη σε αυτήν ε, εξασφαλίζει μία τεχνολογική ηγεσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κινέζοι είναι βασικοί μας ανταγωνιστές και οι Αμερικάνοι και αναγνωρίζουν τον ηγετικό μας ρόλο με συγκεκριμένα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ο τρόπος που συντονιζόμαστε, ο τρόπος που εξασφαλίζουμε την ασφάλειά μας, οι απαντήσεις που δίνουμε στις ε, φυσικές καταστροφές, οι προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές, η αστική και πολιτική προστασία. Όλα αυτά πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα όμως για το διάστημα έχουν πρόβλημα χρηματοδότησης, όπως υπόθηκε και από άλλους. Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο αίτημά μας για χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει επίσης να βρούμε και άλλες μορφές χρηματοδότησης. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι άποψη έχετε για τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εταιρικέ σχέσεις πολυμερούς χαρακτήρα για να ε, εμπλέξουμε καταρχάς και την κοινωνία που την ενδιαφέρουν αυτά τα προγράμματα και για να βρούμε ε, μέσα χρηματοδότησης. Εγώ είμαι πρόεδρος της ε, ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ και ξέρουμε ότι και άλλα κοινοβούλια ε, δουλεύουν ούτω ώστε να δώσουν. Ε, ε, να υπάρχει συνέχεια μετά τη Συμφωνία Κοτονού ε, στην προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ για να προλάβουμε τις φυσικές καταστροφές, τη στήριξη σε πολυμερές επίπεδο, την, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικέ ροές. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα δούμε καλύτερη ε, χρηματοδότηση και τι απάντηση θα έχει η Ευρώπη απέναντι στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα, θα μιλήσει εκ μέρους του ID. Παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή τύχη και εγώ για το Διευθυντή που αποχωρεί και συγχαρητήρια για όλα όσα έκανε, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Για τον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ ιδίω γιατί είχε να κάνει με τα προβλήματα του Γαλιλαίου. Αλλά κατάφερε να ομαλοποίησε και τις σχέσεις ανάμεσα στην GSA και στην ESA. Έγιναν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα που μας επέτρεψαν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ηγετικό ρόλο στον τομέα. Πάνω σε αυτό συμφωνώ και με τον κύριο Σαλίνη, που είναι ο εισηγητής για το πρόγραμμα. Είναι απίστευτο σε ένα τομέα που έδειξε τόσο σημαντική ε, ανάπτυξη και δυναμικό, να σας πω εγώ δηλαδή, ας πούμε για τη δική μου εμπειρία, της μικρής μου, της μικρής και υπανάπτυκτης περιφερειάς μου, που είναι η Απουλία στην, στην Ιταλία, όπου στο διάστημα είμαστε παρόντες από την παραγωγή δορυφόρων σε όλη την αλυσίδα ας πούμε, του διαστήματος η Απουλία συμμετέχει Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, που είναι μία από τις ε, σημαντικές προκλήσεις. Αλλά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχετε καταλάβει πόσες ευκαιρίες μας δίνει αυτή η πρόκληση. Είναι δυσκολία, αλλά ε, είναι και ευκαιρία. Όπως και τα περιβαλλοντικά, ας πούμε. Έχουμε για, τα, για το περιβάλλον, ας πούμε έχουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον εξορθολογισμό των φυσικών πόρων, ε, να τη χρησιμοποιήσουμε για τη γεωργία. Μπορούμε να ελέγξουμε και να παρακολουθήσουμε τη μόλυνση του αέρα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μία, ένας κλάδος ο οποίος έχει μηδενικές εκπομπές. Η... Πρέπει να δούμε το θέμα του προϋπολογισμού. Δεν έχει νόημα να εκφωνούμε λεγίε για όλα όσα έγιναν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά όμως που δεν έγιναν. Εντάξει, υπάρχει τώρα ο κανονισμός, ο οποίος θα προσπαθήσει να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα στη λειτουργία του GSA και ESA. Ε, από την εμπειρία που έχουμε για τη διακυβέρνηση του κοπέρνικου. ίσως το Κοπέρνικος λοιπόν τα πήγε καλύτερα, εντάχθηκε καλύτερα σε σχέση με τον Γαλιλαίο. Ο Κοπέρνικος καλύτερα από τον Γαλιλαίο δηλαδή. Πάντω. εμείς και η Ήτρε έχουμε σωστή στάση. Ο συνομιλητής μας είναι το Συμβούλιο. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τις προκλήσεις ε, και πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή όταν έχουμε αυτόν τον τομέα και που μέσω αυτού του τομέα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις κλιματικές προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην ομάδα ICR και στον κύριο Τσονόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη γλώσσα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμμεριστώ την άποψη του κύριου Σαλίνη και των άλλων συναδέλφων και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εκτελεστικό διευθυντή, κύριο Ντεστορέδας, για το πολύ σημαντικό του έργο. Αυτό που έχετε κάνει στην, στον οργανισμό είναι εκπληκτικό. Είναι τόσο δύσκολο και περίπλοκο το εγχείρημα και εσείς καταφέρατε να το ολοκληρώσετε και να φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο. Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθειά σας. Κανείς δεν θα πίστευε ότι αυτό είναι δυνατόν πριν από πέντε χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνατε πραγματικότητα το 2019. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε αυτή την εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι αυτός ο οργανισμός έχει μεταμορφωθεί σε έναν οργανισμό που ασχολείται με διαστημικά προγράμματα. Έχετε εμπειρία σε πολλά θέματα, πολλούς χώρους, στην ασφάλεια και αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική για άλλα προγράμματα και για το Κοπέρνικος. Είναι ζωτική σημασία η ασφάλεια. Και η ερώτησή μου είναι ίσως όχι τόσο απλή, αλλά είναι έξι. Δεδομένου ότι ο οργανισμός αυτός έχει διευθυνθεί και έχει εκατοντάδες υπαλλήλου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν ε, αρκούν οι εμπειρογνώμονες που έχετε, αν αρκεί το προσωπικό. Αυτοί οι 200 υπάλληλοι που έχετε δεν θεωρώ πως φτάνουν. Ιδιαίτερα δεδομένης της ε, διεύρυνσης ε, του οργανισμού και της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Ο Κοπέρνικος έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι άποψη λοιπόν έχετε γι' αυτό. Κύριε Δεστορέδας, πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον να συντονίσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά προγράμματα, όταν το καθένα από αυτά είναι αρκετά περίπλοκο. Υπάρχουν συνέργειες, αλληλοσυμπληρώνονται τα προγράμματα πώς θα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε. Και μην ξεχνάμε πως ένα από τα σημαντικότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποχωρεί. Τι θα γίνει λοιπόν με το Χαλιλαίο και τα υπόλοιπα προγράμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αποχώρηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα διάφορες εξελίξεις. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε το ανώτερο επίπεδο ποιότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, παίκτης ε, στο, ε, στη τεχνολογία του διαστήματος και θα είναι μεγάλη απώλεια για την Ευρώπη εάν δεν συνεχίσουμε τις καλές σχέσεις με τη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν άλλη μια φορά για το εξαιρετικό σας έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπομπάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσίασή σας και για όλο το έργο που έχετε επιτελέσει. Και εγώ θα κινηθώ στο ίδιο μήκο κύματο ε, με τον συνάδελφο Ντεβέρ. Ε, όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι το πρόγραμμα Γαλιλαίος έχει και μια στρατηγική διάσταση, πολύ σημαντική, τα ερωτήματα λοιπόν που συνδέονται με την ασφάλεια, την αξιοπιστία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει όμως και μια προβληματική ε, που μας προβληματίζει πρόθεσμα, η εύρυθμη λειτουργία των, των διαστημικών προγραμμάτων. Έχουμε ε, πολλά διαστημικά απόβλητα, 8.000 ε, τόνους ε, αποβλήτων λοιπόν ε, που εωρούνται στο διάστημα, τα ξεγνωρίζετε καλύτερα από μένα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος σύγκρουσης αυτών των αντικειμένων με τους δορυφόρους μας, τους δορυφόρους του Γαλιλαίου. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις, κάθε τέτοια σύγκρουση θα οδηγήσει σε περισσότερα ακόμα απόβλητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να αποτρέψουμε αυτές τις συγκρούσεις, να απορριπάνουμε το διάστημα ε, και να αποτρέψουμε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Όλα αυτά υπερβαίνουν βέβαια το πλαίσιο του Γαλιλαίου, αλλά καλό είναι να έχετε μια εικόνα της κατάστασης. Η διαχείριση αυτών των συγκρούσεων, πώς λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Γαλιλαίου. Δεύτερον, Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία για τις τεχνικές ε, λύσεις ε, απορρίπανσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και κατά τη γνώμη σας, δεν έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε ένα διεθνές πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, απορρίπανση του διαστήματος. Και τέλος, η μείωση των διαστημικών αποβλήτων έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των δορυφόρων ε, που χρησιμοποιούνται σήμερα στο Γαλιλαίο. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις και σας ευχαριστώ και για το έργο που έχετε επιτελέσει. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Να πω και εγώ δύο λόγια. Γενικά για το διάστημα και για τον οργανισμό σας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ιδίω ε, ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα και την ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων μας. Πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Θεωρώ επίσης ότι στα διαστημικά μας προγράμματα μπορούμε να βρούμε ακόμα και απαντήσεις για την επίτευξη των στρατηγικών μας ε, στόχων που συνδέονται με την Πράσινη Συμφωνία, για παράδειγμα απομάκρυνση από τον άνθρακα, ενεργειακή απόδοση, οικονομία με γνώμονα ε, την καινοτομία μέχρι το 2050. Πολλά από αυτά που κάνετε και εσείς και άλλοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των ε, στόχων και στη βελτίωση της οικονομίας μας. Επιπλέον θα πρέπει να κατοχυρώσουμε την απαραίτητη ε, χρηματοδότηση και σωστά είπαν οι συνάδελφοι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη και τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ανταγωνισμό στο διάστημα, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς. Και εδώ θα πρέπει να υπερασπιστούμε τουλάχιστον την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ε, κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να έχουν ακόμα παραπάνω. Αυτό προτείνει το Κοινοβούλιο. Αλλά αν υπάρξει περικοπή 10%, 10,7% του διαστημικού προγράμματος, τότε ακόμα και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, όπως ε, το πρόγραμμα Γαλιλαίος και Κοπέρνικους, θα πιεστούν. Και θα είναι σίγουρα δύσκολο να δημιουργήσουμε και νέα προγράμματα. Μετά, οι συνέργειες με το Ταμείο Άμυνας και το ερευνητικό μας πρόγραμμα, Horizon Europe. Υπάρχουν εδώ δυνατότητες, ευκαιρίες για τη διαστημική έρευνα και τα προγράμματά σας. Έχετε λοιπόν τη στήριξή μας. Η Επιτροπή μας είναι καθήλυνα αρμόδια σε ό,τι αφορά τις ε, διαστημικές δραστηριότητες και τη διαστημική πολιτική και είμαστε καθόλου έτοιμοι να σας στηρίξουμε μαζί και με άλλα εμπλεκόμενα μέρη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια, για το διάστημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήματα, να προσθέσετε ενδεχομένως άλλες ε, παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα τηρήσω το δεκάλεπτο που μου αναφέρατε και προηγουμένως. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, ε, γιατί πολλές φορές ε, θίξατε παρόμοια ζητήματα. Ξεκινώ από το ζήτημα του προπολογισμού. Πολλοί από εσάς ε, ανέφεραν το θέμα αυτό και ότι θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να εισακουστεί το αίτημά σας ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι το διαστημικό πρόγραμμα και ο προπολογισμό ε, έχουν ένα αυστηρό πλαίσιο. Δεν γίνεται να έχουμε ένα σύστημα γαλλιλαίος με 20 δορυφόρους, γιατί δεν θα έχουμε τη σωστή απόδοση. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τις απαιτήσεις του συστήματος. Μια περικοπή του προπολογισμού αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε ελλείψεις και αδυναμίες που θα έπληταν την επιτυχία του συστήματος. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος, επίσης, γιατί ε, μια περικοπή του προπολογισμού θα ε, μπορούσε να αποβεί σε βάρος ε, του κατάντη τομέα. Να σας υπενθυμίσω ότι εκεί έγκυται και μεγάλο κομμάτι της αξίας του προγράμματος. Η Ευρώπη πραγματικά θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό το σκέλος. Ο οργανισμός μας που ασχολείται με αυτόν τον προπολογισμό ε, προτείνει αύξηση και τριπλασιασμό μάλιστα του προπολογισμού σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. αναμένουμε έναν προπολογισμό περίπου στα 700 με 750 εκατομμύρια κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της επταετίας. Αν δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία στις ΗΠΑ, ε, πραγματικά δεν υπάρχει σύγκριση. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι σημαντικό και το ποσό το ύψος του προπολογισμού, αλλά και ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί. Μπορώ να σας πω ότι πρόσφατα, για παράδειγμα, υπογράψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές ιδέες, προτάσεις και πρωτοβουλίες που μπορούμε να προωθήσουμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με νέους ε, παράγοντες της αγοράς. Με τα χαράς άκουσα το ερώτημα του κυρίου Τεσενόφσκι για τον προπολογισμό του οργανισμού. Γιατί γίνεται λόγος για τον προπολογισμό των προγραμμάτων, αλλά και ο ίδιος οργανισμός, ο GSA, περνάει δύσκολες μέρες. Γιατί υπάρχει υποτίμηση του βασικού προπολογισμού που απαιτείται για την ε, λειτουργία του οργανισμού. Και σας παροτρύνω να δείτε ένα ενδιαφέρον έγγραφο ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018. Θα το βρείτε στον ιστότοπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, ο οργανισμός μας είναι μεσαίου μεγέθους από πλευράς προσωπικού. Αλλά αν δείτε τον προπολογισμό, τα έσοδα, έχουμε τρομερά αποτελέσματα. Αυτό σας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα στον προπολογισμό και το προσωπικό μας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τον προπολογισμό των προγραμμάτων, αλλά και τον προπολογισμό του οργανισμού. Πράγματι, Το Γαλιλαίο εξετάζει πολλούς ε, διαφορετικούς ε, τομείς. Σίγουρα η Πράσινη Συμφωνία είναι ένας τομέας ενδιαφέροντος. Μπορώ να σας δώσω πολλά στοιχεία από την ανάλυση μας που δείχνουν την ε, εξοικονόμηση, την μείωση των εκπομπών διεξοδίου του άνθρακα, την εξοικονόμηση καυσίμων, ε, τη μείωση της χρήσης ζυζανιοκτώνων που προκύπτουν ακριβώς από την χρήση του Γαλιλαίου και του Έγνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, χρήση, τη λειτουργία του συστήματος και την ε, δυσκολία προσλήψεων, βελτιώνεται η κατάσταση με τα χρόνια, στην αρχή υπήρχε σοβαρή δυσκολία. Αλλά όλο και περισσότερο γίνεται διαχειρίσιμο το ζήτημα. Γιατί και εμείς λαμβάνουμε μεγαλύτερη προβολή, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, τον οργανισμό και αυτό αντανακλάται και στην δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού. Κάποιοι ρώτησαν ε, για τα διαστημικά απόβλητα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ε, μπορεί να έχετε ακούσει για ε, μια συστοιχία χιλιάδων δορυφορών Μας απασχολεί λοιπόν όλο ένα και περισσότερο. Για το Γαλιλαίο βρισκόμαστε σε σχετικά καλή κατάσταση. Γιατί χρησιμοποιεί δορυφόρους με μια τροχιά 22.000 χιλιόμετρων από ε, την γη. Υψηλή τροχιά λοιπόν σχετικά, επομένω το πρόβλημα είναι λιγότερο σοβαρό. Σήμερα διαχειριζόμαστε αυτόν τον κίνδυνο με υφιστάμενα προγράμματα παρακολούθησης άλλων χωρών, κυρίως τον είπα. που παρακολουθούν τα αποβλήματα τα απόβλητα και σε ε, περίπτωση σύγκρουσης ε, αυτό θα μας επέτρεπε να ε, μετακινήσουμε τους δορυφόρους σε διαφορετική τροχιά και έτσι να αποτρέψουμε τον κίνδυνο. Αλλά είναι απαραίτητο και για την Ευρώπη να αποκτήσει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Το είπα και πριν, προγράμματα όπως ε, ε, το σύστημα διαχείρισης ε, διαστημικής κυκλοφορίας, διακίνησης. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε τις εξελίξεις για να είμαστε και σε θέση να διαχειριστούμε αυτό το αναδυόμενο ζήτημα. Άλλη ερώτηση αφορούσε λοιπές ε, πηγές χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Συνήθως ε, απαντώ ότι η Ευρώπη με τον Γαλιλαίο και το Έγνος ε, δημιουργεί υποδομές, σαν να φτιάχνουμε έναν αυτοκινητόδρομο. Και αναμένει ότι θα έχει απόσβεση αυτής της επένδυσης ε, με ωφέλη στην οικονομία, όπως γίνεται και στα υπόλοιπα έργα αποδομών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορούμε να δούμε την σύζευξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ, στον τομέα κατά αντί πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κέντρων αριστείας, για να φτάσει το διαστημικό πρόγραμμα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη με τις επενδύσεις που γίνονται σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κλάδου, σε βιομηχανικό επίπεδο. Αντί να έχουμε τρεις-τέσσερις χώρες που επενδύουν ε, στη γεωργία ακριβίας, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα-δύο τέτοια κέντρα και άλλες χώρες ε, να ασχολούνται με τα αυτόνομα οχήματα, ε, με τη σηματοδότηση των σιδηροδρόμων και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο εξορθολογισμού των επενδύσεων και αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Κάτι τελευταίο για το Brexit. Ναι, είναι λυπηρό που θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη και για το διάστημα και για τον Γαλιλαίο πιο συγκεκριμένα και το έγνος. Ήταν από τους ε, βασικούς εταίρους μας αυτό το θέμα. Βέβαια αυτό αφορά περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά από πλευράς μου μπορώ να σας πω ότι πραγματικά θα ήθελα μια συμφωνία όπως έχουμε σήμερα. Όπως, με χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία. Οι χώρες αυτές συνεισφέρουν ένα μερίδιο του ΟΑΕΠ τους ε, στο πρόγραμμα και φυσικά έχουν και τα πλήρη ωφέλη της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Για την ασφάλεια βέβαια πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διευθετήσεις, αλλά σίγουρα θα βρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τεστορίδες που ήρθατε και μας μιλήσατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την πολύτιμη εισφορά σας σε αυτήν την ε, συζήτηση. Σύντομα θα ακολουθήσει και η ανταλλαγή απόψεων με τον άλλο οργανισμό, τον ΕΙΣΑ. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε, όμως ε, θα γίνει σύντομα. Δυστυχώς σήμερα ο διευθυντή ε, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος δεν μπορούσε να έρθει. Θα ολοκληρώσω την πρωινή συνεδρίαση σε αυτό το σημείο. Μην ξεχνάτε όμως ότι πρέπει να γυρίσουμε μία ώρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, διότι θα γίνει ανταλλαγή απόψε με την ε, Επίτροπο Βεστάρα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ.